Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Δεν έχει ζητήσει μέχρι τώρα κάποιος ε, να αλλάξει κάτι στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Πριν ξεκινήσουμε τις κανονικές μας εργασίες, ο κύριος Οντί έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι στην ερμηνεία του 191, του άρθρου 191, μιας και δεν υπήρξε διαφορετική άποψη για την ερμηνεία αυτή, για τη